γράψαμε το 2009 Συμφωνία Σύνδεσης και Συνεργασίας και με μεγάλη ευχαρίστηση καλωσορίζω εδώ πέρα τους Ινδονήσιους βουλευτές. Επόμενο θέμα, προς ενημέρωση. Ο κύριος Μάικ Νάτρας έφυγε από το κόμμα της Ευρώπης για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία και από τις 23 Ιουνίου 2010 θα λογίζεται με τους μη εγγεγραμμένους. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές